Mes Αγαπητοί συνάδελφοι, καλησπέρα σας. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε τη συνεδρίασή μας. Λοιπόν, κύριε Βίβαντενκάμπ, βγάλτε το σακάκι και καθίστε για να ξεκινήσουμε. Το σακάκι μόνο βγάλτε. Λοιπόν, μπορούμε να εγκρίνουμε την ημερήσια διάταξη. Θεωρώ πως ναι, αν δεν υπάρχουν αντιρρήσεις, Ανακοινώσεις της Προέδρου. Δεν έχω ανακοινώσεις, επομένως μπορούμε ευθύς αμέσως να περάσουμε στο σημείο 3 που αφορά την πολιτική συνοχή και το θεματικό στόχο για την προαγωγή των βιώσιμων μεταφορών και την εξάλληψη των σημείων συμφόρενσης στις υποδομές των βασικών δικτύων. Η συγκεκριτή είναι ο κύριος Σλοτόφσκι. Κύριε Σλοτόφσκι θα σας δώσω το λόγο και εν συνεχεία θα ακούσουμε τους κοιόδης εισηγητές και βέβαια όλα τα υπόλοιπα μέλη της Επιτροπής που επιθυμούν να πάρουν το λόγο και στο τέλος θα ζητήσω από τον ή την εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να πάρει το λόγο. Πάντως δίνω καταρχάς το λόγο σε εσά κύριε Σλοτόφσκι και σας καλημερίζω. Καλημέρα σας κύριε Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ πολύ που μου δίνετε το λόγο Χαίρομαι πάρα πολύ που μπορώ να ξεκινήσω τις εργασίες μας για ένα πολύ σημαντικό θέμα όσον αφορά αυτή την περίοδο προγραμματισμού για την προαγωγή των βιώσιμων μεταφορών και την εξάλληψη των σημείων συμφόρησης στις υποδομές των βασικών δικτύων. Πρέπει εμείς να συντάξουμε μια γνωμοδότηση για την Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης και ξέρετε ότι ε, στα πλαίσια του περιορισμένου κειμένου που μας επιτρέπεται στα πλαίσια μιας γνωμοδότησης δεν μπορούμε να καλύψουμε πάρα πολλά πράγματα. Δεν θα ήθελα να επισέλθω σε πάρα πολλές λεπτομέρειες. Πάντως είναι πάρα πολύ σημαντικό να τονίσουμε ότι τόσο το Ταμείο Συνοχής όσο και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης όσο και ο μηχανισμός συνδεοντα την Ευρώπη είναι οι βασικοί μηχανισμοί χρηματοδότησης όσον αφορά τις υποδομές μεταφορών. Αυτό δεν θα πρέπει να τροποποιηθεί στο μέλλον. Περίπου 70 δισεκατομμύρια ευρώ έχουν δεσμευθεί για την περίοδο 2014-2020 20 και 45 δισεκατομμύρια από το Ταμείο Συνοχής και 40 περίπου δισεκατομμύρια από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης. Θα μπορούσε κανείς να αναρωτηθεί αν η θεματική συγκέντρωση έχει όντως υποστηρίξει τον τομέα των μεταφορών, ο τομέα των μεταφορών συμβάλλει πάρα πολύ στην οικονομική ανάπτυξη της Ευρώπης και στην ανταγωνιστικότητα των περιφερειών μας. Αυτό το οποίο χρειάζονται οι περιφερειές μας είναι καλύτερες υποδομές μεταφορών προκειμένου να καταφέρουν να τονώσουν περισσότερο την οικονομική του ανάπτυξη, προκειμένου να προωθήσουν περισσότερο την ενιαία αγορά, καθώ επίση και την οικονομική και δαφική συνοχή. Ο προγραμματισμός στα πλαίσια της θεματικής κέντρωσης δεν έχει τροποποιηθεί πολύ. Η πρόοδος όσον αφορά όμως τα διευρωπαϊκά δίκτυα μεταφορών ήταν αρκετά περιορισμένη τελευταία. Τα δεδομένα τα οποία μας δίνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καταδεικνύουν ότι η κατάσταση είναι κάπως τρομακτική. Βλέπουμε ότι υπάρχει ένα πολύ χαμηλό επίπεδο απορρόφησης των ε, κονδυλίων τα οποία εκταμιεύονται για να γίνουν οι απαραίτητες επενδύσεις. από τα 9.600 χιλιόμετρα που προγραμματίζονταν προς κατασκευή όσον αφορά την οδοπία, μόνο τα 1.900 χιλιόμετρα έχουν πραγματοποιηθεί. Τα στατιστικά δεδομένα επίσης είναι ακόμα πιο ανησυχητικά. Από τα προγραμματισμένα 700 χιλιόμετρα σιδηροδρομικών χιλιόμετρων, μόνο 982 χιλιόμετρα έχουν πραγματοποιηθεί, ενώ 16 μόνο χιλιόμετρα αφορούν τις διασυνδέσεις τις δρομικές και τις οδικές που έπρεπε να είχαν πραγματοποιηθεί. Ο αρχικός στόχος ήταν πολύ υψηλότερο. Από το 2007 έως το 2013 επενδύσαμε 81 δισεκατομμύρια ευρώ. Περίπου το 1 τρίτο μόνο των συνολικών διαφορετικών ταμείων για τις επενδύσεις. Δεν νομίζω ότι θα πρέπει να απολέσουμε τα υπόλοιπα κονδύλια τα οποία ακόμα εκκρεμούν προς επένδυση. Έχουμε πει ότι από το 2015 και μετά ο τομέας των μεταφορών θα αυξηθεί κατά περίπου 50%. Πολλά κράτη-μέλη όμως φαίνεται ότι υπολείπονται ακόμα σε σχέση με την πραγματοποίηση των κοινών στόχων στον τομέα των μεταφορών, ιδίω αν συγκρίνουμε τη Δυτική Ευρώπη με τις κεντρικές και χώρε χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εδώ πέρα βλέπουμε ότι οι επενδυτικέ προτεραιότητες τη Ευρωπαϊκής Ένωσης συχνά δεν συνάδουν με τις πραγματικές ανάγκες των λιγότερων απτυγμένων κρατών μελών τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Γι' αυτό το λόγο ζητώ από όλους μας να επιδείξουμε ευελιξία κατά τη χρηματοδότηση των έργων προκειμένου να γεφεριωθεί το κενό αυτό το χάσμα που υπάρχει σε επενδύσεις. Πρέπει επίσης να πούμε ότι τα κράτη-μέλη πολύ συχνά δεν καταφέρνουν να διαχειριστούν σωστά τα διαφορετικά κονδύλια, τα διαφορετικά μέσα χρηματοδότηση τα οποία εφίστανται για τον τομέα των μεταφορών. Πρέπει λοιπόν να ενημερώσουμε καλύτερα τα κράτη-μέλη σε σχέση με τα εφιστάμενα μέσα χρηματοδότησης. Και ξέρετε ότι πολύ συχνά τα μικρά κράτη-μέλη ε, αντιμετωπίζουν δυσκολίες κατά την ολοποίηση των συμπράξεων δημοσίου διωτικού τομέα. Συνεπώς, θα πρέπει να ενισχυθεί το σκέλος επιχορηγήσεων των πόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να μην βασιζόμαστε μόνο στα χρηματοδοτικά μέσα. Τα χρηματοδοτικά μέσα τα οποία υφίστανται αυτή τη στιγμή δεν είναι τα πλέον κατάλληλα πολλές φορές όσον αφορά τις επενδύσεις πρέπει να γίνουν στις οδικές, στις μεταφορές, στις εσωτερικές πρώτες οδούς κτλ. Τονίζω ότι θα πρέπει να διατηρήσουμε τις επιχορηγήσεις γιατί μόνο μέσω επιχορηγήσεων από την Ευρωπαϊκή Ένωση θα καταφέρουμε να προσελκύσουμε και ιδιωτικά κεφάλαια. Θα πρέπει επίσης να γίνουν και απαραίτητε προσαρμογές στο νέο πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση να μειωθεί στο νέο αυτοπλαίσιο χρηματοδότηση για το μέτρο μεταφορών. Τα κονδύλια εξακολουθούν και ιδιαίτερα σημαντικά προκειμένου να δημιουργήσουμε έναν ενιαίο ευρωπαϊκό χώρο μεταφορών. Α μην ξεχνάμε ότι τα κράτη-μέλη αντιμετωπίζουν κοινέ προκλήσει όσον αφορά τη χρηματοδότηση τη υποδομή των μεταφορών και πολλέ φορέ αναγκάζονται να λειτουργήσουν με πολύ περιορισμένου εθνικού προπολογισμού η μερίδα του λέοντος για την χρηματοδότηση των ε, έργων μεταφορών εξακολουθεί και επιβαρύνει τα κράτη-μέλη. Ας μην το ξεχνάμε αυτό. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κυρία Σλοτόφσκι. Αρχίζει η συζήτηση. Οι σκιώδεις έχουν το λόγο. Ο κύριος Βιμ Βαντεκάμπ έχει το λόγο. Κυρία Πρόεδρε, σας ευχαριστώ. και έχω την τιμή να αντικαθιστώ τον συνάδελφο Μαριάν Μαρινέσκου σήμερα το απόγευμα, ο οποίο είναι σκιώδη εισηγητής από την ομάδα του ΕΛΚ. Για τον συνάδελφο του ECR θα ήθελα να κάνω τρει παρατηρήσει. Ε, πρώτη παρατήρηση. Οι τρεις ερωτήσεις που θα θέσω ουσιαστικά περιλαμβάνονται στην ε, έκθεση του κυρίου Σλοτόφσκη. Το θέμα λοιπόν είναι όντως ε, η υλοποίηση των ε, διαδρόμων T. Η υλοποίηση των διαδρόμων αυτών. Γιατί συχνά τα κράτη-μέλη μένουν πίσω. Μένουν πίσω στην οργάνωση, στη συγχρηματοδότηση των διαδρόμων. Έχουμε την αρχή του use it or lose it. Ε, της χρήσης δηλαδή, των πόρων ή απώλειας αυτών. Δεν ξέρω αν ο κύριος Σλουτόφσκι θα ήθελε να πει δύο λόγια γι' αυτό. Τώρα, δεύτερη ερώτηση για το ESF. Το είπε πολύ ευγενικά, αλλά φυσικά όλοι βρισκόμαστε στη, φάμεση, στη φάση διαπραγματεύσεων αναπίσημα και επίσημα για το νέο πουδουπού ή επάση περιπτώσει για την συνέχεια των πόρων του ESF, τον, του ΣΕΦ μάλλον, των ε, κονδυλίων ΣΕΦΕ. για το Connective Europe Facility και τους πόρους του. Αν θα θέλετε να σχολιάσετε και τέλος να μας πείτε τη λόγια για τις γειτονικέ χώρες. Βλέπουμε την προσέγγιση της κυρίας Μπούλς αλλά και την κυρίου Χάν. Διαπιστώνουμε ότι συχνά θέλουμε να τραβήξουμε γραμμές από την Πολωνία στην Ουκρανία, από την Τσεχία, στη Ρουμανία, στη Μολδαβία. Το ερώτημα λοιπόν είναι κατά πόσο το στοιχείο αυτό θα μπορούσε να συμπεριληφθεί και αυτό στο σχέδιο γνωμοδότηση, γιατί οι δρόμοι μα ασφαλώ δεν σταματούν στα εξωτερικά σύνορα τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ τον κύριο Βιμ Βαντεκάμπ. Εντάξει, πιείτε και λίγο νεράκι. Ο κύριος Έρτουγκ. Η κυρία Γκραπίνη τότε. Ουδής. Ο κύριος Τελίτσκα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα μιλήσω εξ ονόματος του κυρίου Μίλτεμπουργκ και σκέφτηκα να μιλήσω Ολλανδικά. Τον αντικαθιστώ γιατί είναι ε, άρρωστος και δυστυχώς δεν μπόρεσε να παρευρεθεί. Εξ ονόματος του θα ήθελα να πω ότι καλωσορίζει τη γνωμοδότηση και όπως ε, και άλλοι συνάδελφοι έχει ορισμένα σχόλια θα πρέπει να ανοίξουν οι δυνατότητες για να χρησιμοποιηθεί το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής για τις ε, διασυνοριακές εργασίες υποδομής και επίσης τα μικρότερα σχέδια, τα ε, διασυνοριακά, θα πρέπει να τύχουν υποστήριξης. Θα πρέπει να υπάρχει συμμόρφωση με ερεσιμότητες εξάντε και το τελευταίο σχόλιο αφορά την παράγραφο 4 θεωρεί ότι αυτές οι επιχορηγήσεις θα πρέπει να αυξηθούν μέσα στα πλαίσια της συνέργειας ιδιωτικού και δημόσιου τομέα και ε, φυσικά και μέσα στα πλαίσια της κρατικής συνδρομής. Αυτά έχω να πω από τον συνάδελφο. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Τελίτσκα. Ο κύριος Πιμέντα Λόπες έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Έχουμε ορισμένες αποκλήσεις σε σχέση με την άποψη της ε, Ρέτζη όταν προσπαθούμε να κάνουμε μία διασταύρωση μεταξύ αναγκών και πολιτικών συνοχής και της παρουσίασης της ενιαίας αγοράς που είναι ένα βασικό μέσο για να φτάσουμε στους ε, απότερους στόχους οι οποίοι ορίζονται από την πολιτική συνοχής. Αντίθετα, βλέπουμε ότι οι ίδιοι κανόνες της αγοράς έχουν επιβάλει συρρυκνώσεις έτσι ώστε να μην εμβαθύνουμε την συνοχή αλλά τη δυσαναλογία μεταξύ κρατών μελών ιδιαίτερα και στον τομέα των μεταφορών. Άρα δεν μας εκπλήσει το γεγονός ότι η ίδια στρατηγική που οδήγησε σε ιδιωτικοποιήσεις σε ολόκληρη την Ευρώπη ορίζεται με βάση αυτά τα δύο έγγραφα. Γι' αυτό η το στρατηγικό όραμα για τον τομέα ε, βρίσκεται εκτός ε, δημόσιου τομέα όπως θα έπρεπε. Και γι' αυτό δεν μας εκπλήσει και το γεγονός ότι υπάρχει έλλειψη αναφοράς ε, του δημοσίου τομέα και δυστυχώς ο δημόσιος τομέας αναφέρεται πενιχρά στα δύο ε, έγγραφα όταν μιλάμε για την ε, σύνδεση, συνοχή ιδιωτικού και δημόσιου τομέα και τη συνέργεια των δύο τομέων. Γιατί πέρα από το υψηλό οικονομικό κόστος για τα κράτη-μέλη υπάρχει και ένα αντίτιμο που πληρώνουν οι πολίτες. Δηλαδή βλέπουμε αύξηση του κόστους και μείωση της, πυρό... της ποιότητας παροχής υπηρεσιών. Μιλάμε δηλαδή για άση των περιορισμών στην κυκλοφορία, στα οδικά και σιδηροδρομικά δίκτυα και αυτό μπορώ να πω ότι ισχύει στη χώρα από την οποία προέρχομαι, την ε, Πορτογαλία, διότι το οδικό ε, δίκτυο εκχωρείται σε ιδιωτικό τομέα μέσα στα πλαίσια αυτής της συνέργειας ε, ιδιωτικού και δημόσιου τομέα και γι' αυτό ε, σε τελευταία ανάλυση η όλη εκχώρηση γίνεται προς τον ιδιωτικό τομέα. Άρα τα πράγματα διαφέρουν από την άποψη του εγγράφου Θεωρούμε ότι ο δημόσιος τομέας θα πρέπει να υπηρετεί τις κοινέ μεταφορές καθώς και τις ε, υποδομές έτσι ώστε να υποστηριχθούν οι μακροοικονομικές πολιτικές σε κάθε κράτος μέλος. Ευχαριστούμε. Ο κύριος Κράμερ έχει το λόγο. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε και να ευχαριστήσω ασφαλώς και τον εισηγητή για την γνωμοδότηση και για την παρουσίαση. Προφανώς το θέμα αυτό είναι βασικό η περιφερειακή ανάπτυξη της Ευρώπης. Και μαζί με την Επιτροπή των Περιφερειών ε, έχουμε καλή συνεργασία από την Επιτροπή μας και καταφέραμε να περάσουμε να ασχοληθεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με το θέμα των διαστοριακών αυτών δικτύων. Μιλάμε για δισεκατομμύρια ευρώ τα οποία δαπανώνται, για παράδειγμα, στα συνδροδρόμους. Αλλά είναι κατακριμονισμένη ακόμα η κατάσταση. Με την τελευταία λοιπόν πρόταση που αναφέρεται ότι θα πρέπει τα κράτη-μέλη να ε, δραστηριοποιηθούν. Εδώ είναι το ζουμί, γιατί θεωρώ ότι τα κράτη-μέλη δεν κοιτούν την ε, ευρωπαϊκή υπεραξία. Κοιτάνε μόνο τα εθνικά του συμφέροντα. Αυτή είναι η εμπειρία η δική μας. Γι' αυτό λοιπόν είναι θετικό και σημαντικό το γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να διαθέσει πλέον τα 117 εκατομμύρια για τις συνοριακές αυτές ε, ε, συνδέσεις. Τα κράτη-μέλη. Από το Μόναχο στο Βερολίνο, ένα παράδειγμα να σας δώσω, να σας πω ότι η απόσταση πλέον είναι δύο ε, ώρες λιγότερες. Ε, δέκα δις κόστησε αυτό και 500 εκατομμύρια συνέβαλε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά έχουμε 50 χιλιόμετρα, ε, κενό μεταξύ Πολωνικής πόλης και Κόμπλεντσε. Και αυτό μπορούμε λοιπόν να το κλείσουμε το κενό και να ε, μειώσουμε την απόσταση στο τρένο κατά δυόμιση ώρες ε, είναι μικρό ποσό σε σχέση με το συνολικό ποσό αλλά κανείς δεν θέλει να το δώσει η Γερμανία λοιπόν δήλωσε το πρόγραμμα αυτό είχαν διευκρινιστεί τα πάντα η χρηματοδότηση είχε οργανωθεί σε εθνικό επίπεδο και διαπίστωσαν στη συνέχεια ότι υπάρχουν και ευρωπαϊκοί πόροι για να κάνουν, και ζήτησαν λοιπόν του ευρωπαϊκού αυτού πόρου για να κάνουν το ίδιο. Θα ήθελα λοιπόν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ε, έλεγε ότι κοιτάξτε, κλείστε και αυτό το κενό πια μεταξύ Κόμπλεντς και Πολωνικών συνόρων. Ε, να σας δώσουμε την χρηματοδότηση, αλλά φροντίστε και την ευρωπαϊκή πραξία. Δεύτερο θέμα. Το θέμα της διαλειτουργικότητας θα πρέπει να το φροντίσουμε και εδώ θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να είναι πιο α, αυστηρή. Είπατε ότι υπάρχουν περιοχές δεκάδες χιλιάδες χιλιόμετρα τα οποία δεν έχουν σιδηροδρόμους. Και εδώ λοιπόν θα πρέπει να υπάρξει ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία. Και τελευταίο θέμα που ήθελα να αναφέρω είναι το εξή. Αντίθετα με τα εθνικά κράτη έχουμε τι ευρωπαϊκέ ε, διαδρομέ. Έχουμε δηλαδή ευρωπαϊκή αρμοδιότητα σε ό,τι αφορά τα ποδήλατα. Ξέρετε ότι είμαι μεγάλο συμπαρμαχό των ποδήλατων και εδώ υπάρχουν λοιπόν ευρωπαϊκοί πόροι και αυτό θα πρέπει να λεφθεί υπόψη. Ένα μικρό ποσοστό τουλάχιστον να δαπανάτε και για τους ποδηλατοδρόμους που προωθούν και τον τουρισμό με ποδήλατο. Αυτό προωθεί συγκεκριμένες περιοχές και την τελευταία εβδομάδα ενημερώθηκα για ένα αριθμητικό στοιχείο στο Ροδεμβούργο, στη Γερμανία. 23% όλου του τουρισμού είναι ποδηλατικός τουρισμός. Έχει και οικονομικές επιπτώσεις λοιπόν ο τουρισμός αυτός και θα έπρεπε να ληφθεί ενδεχομένω υπόψη πιο πολύ. Πιο πολλά χρήματα. Όχι απαραίτητα θα έλεγα. Δεν χρειαζόμαστε πιο πολλούς πόρους. Όχι. Διαφορετική πολιτική χρειαζόμαστε. Γιατί αν συνεχίσουμε ως, όπως ως τώρα και κοιτάμε τα μεγάλα προγράμματα που έχουν ξεκινήσει πριν από 20-30 χρόνια δεν θα βγάλουμε άκρη. Η ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία θα πρέπει να αποτελεί τη μεγαλύτερη προτεραιότητα για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και θα ήθελα λοιπόν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να παρέμβει πιο ενεργά. Υπάρχει περιορισμό λοιπόν των ε, πόρων και προς την κατεύθυνση αυτή θα πρέπει να κινηθούμε. Ευχαριστώ. Ε, ευχαριστώ. Ε, ο κύριος Ο κύριος έχει το λόγο. Θα είμαι πολύ σύντομος. Ήθελα απλώς να πω ότι δεν μετράει μόνο ο όγκος και θεωρώ ότι θα πρέπει να κρατήσουμε τις γραμμές του προϋπολογισμού. Αυτό όμως που έχει σημασία είναι προς τα που κινούνται αυτοί οι πόροι, αυτά τα κονδύλια. Έχετε ένα σαφές παράδειγμα, δηλαδή στις πολιτικές ανταγωνισμού και συνοχής, η ανταγωνιστικότητα δεν, ε, μάλλον ε, ο τομέας των μεταφορών δεν έχει πρόσβαση στον ανταγωνισμό. Κάτι τέτοιο απαγορεύεται. Επίσης, όταν μιλάμε για πολιτικές συνοχής, τότε υπάρχει μεγάλη διάχυση. Δεν μπορούμε να ζητήσουμε ένα προϊόν υψηλής προστιθέμενης αξίας και μετά να το εγκαταλείψουμε, διότι ε, τα σχέδια στον τομέα των μεταφορών όταν έχουν μεγάλη προστιθέμενη αξία πολλές φορές δεν συμβαδίζουν με τους στόχους μας. Όταν λοιπόν έχετε να κάνετε με μία εκδήλωση ενδιαφέροντος, έχετε ποσοτικά και ποιοτικά στοιχεία που δεν συνάδουν με την ε, πολιτική συνοχής. Έμπρακτα λοιπόν όλα εξαρτώνται από την ποσότητα αλλά και τη διαχείριση. Και το πρόβλημα της πολιτικής συνοχής είναι ότι υπάρχει διάχυση και όχι συγκέντρωση, γι' αυτό δεν θα έχουμε ευρωπαϊκά σχέδια τη θέμενης αξίας. Υπάρχουν 11 δις που μπήκαν από την συνοχή στο ΣΕΦ. Βλέπετε όμως ότι αυτά τα 11 δις ε, τα πήγαν πολύ καλύτερα από ολόκληρο το τομέα της συνοχής τα 6 προηγούμενα χρόνια. Ναι, χρειάζονται χρήματα, αλλά χρειάζεται και καλή διαχείρισή τους. Όταν βλέπουμε τα αποτελέσματα διαπιστώνουμε ότι όταν υπάρχει καλή διαχείριση έχουμε και πολύ καλά αποτελέσματα, ενώ όταν υπάρχει κάκο διαχείριση το αντίθετο. Τώρα στρέφομαι προς την Επίτροπη και θα δώσω το λόγο στον κύριο Βενσάν Λίνερ από τη Γενική Διεύθυνση Ρίτζιο. Σας ευχαριστώ πολύ που δίνετε το λόγο και έχουμε δύο σημεία στα οποία θα θέλαμε να σχολιάσουμε. Καταρχά συντομία. Καταρχάς την παράγραφο D, η, ε, η οποία αναφέρει τα ποσά που μεταφέρονται στο ERDF από τους ευρωπαϊκούς πόρους μέσω των σχετικών προγραμμάτων. Εδώ στην παράγραφο D θα θέλαμε να υπάρξει ε, αναφορά στην ΣΕΦ, στο Connective Euro Facility ε, και σε ό,τι αφορά τα επιπλέον ποσά που διατίθενται μέσω του ΣΕΦ στο επίπεδο 1,3 δις που έχουμε από τα Ταμεία Συνοχής και από το Γενικό Φάκελο. το δεύτερο, έχουμε αμφιβολίες στην παράγραφο 1 σε ό,τι αφορά την αναφορά που γίνεται σε πολύ χαμηλό ποσοστό επιλογής έργων. Εδώ έχουμε πρόσφατα στοιχεία από την έκθεση του Ιανουαρίου σε ό,τι αφορά την υλοποίηση των Ταμείων Συνοχής στο ERDF με ημερομηνία καταληκτική 2017. Τα στοιχεία που έχουμε είναι ότι είμαστε πάνω στο 61,5% σε ό,τι αφορά τα ποσοστά επιλογής, σε ό,τι αφορά το TNT, είμαστε στο 64% ποσοστό επιλογής και κοιτώντας ε, στους σιδηροδρόμους τα σχετικά προγράμματα, είμαστε στο 66% σε ποσοστό επιλογής έργων. Και σε ό,τι αφορά την πολιτική συνοχή, ο αριθμός ε, είναι επίσης ε, πολύ υποσχόμενος μετά από τέσσερα χρόνια έναρξης της περίοδου. Μεγάλο ποσοστό του προπολογισμού έχει ήδη εκχωρηθεί σε προγράμματα. Τα δεδομένα αυτά χορηγήθηκαν και στο σχέδιο γνωματοδότηση τη Επιτροπή Περιφερειακή ανάπτυξη για τα χιλιόμετρα των επιλεγμένων προγραμμάτων. Αυτά είναι στοιχεία τα οποία συλλέξαμε το Μάιο 2017 με την ημερομηνία καταρακτική 2016. Έξω έχουν υπάρξει πολλές εξελίξεις, υπάρχουν δύο μηχανισμοί. Η πρώτος είναι ότι μέχρι το τέλος του 2016 η προστασία των εθνικών εχωρήσεων, στα πλαίσια του Connective Euro Facilities ε, τερματίστηκε και έτσι εστιαστήκαμε πιο πολύ στα ε, προγράμματα συνοχή και η περίοδος 2007-2013 ολοκληρώθηκε κοιτώντα επίσης τα τελευταία δεδομένα και πάλι η επιλεξιμότητα, η επιλογή προγραμμάτων είναι πολύ θετική. Σας ευχαριστούμε πολύ. Να ξαναδώσω τώρα το λόγο στον εισηγητή, τον κύριο Σλοτόφσκι. Έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, συμφωνώ, συμφωνώ με τις παρατηρήσεις σας μετά σου υπόθηκαν ε, κατά τη διάρκεια της συζήτησης αυτής. Ελπίζω ότι θα καταθέσετε και καλές τροπολογίες, έτσι ώστε να τις ενσωματώσω εν συνεχεία στη γνωμοδότηση αυτή. Θα θέλα να αναφερθώ σε αυτά τα οποία είπε ο κύριος Βάντεν Κάμπ. Όσον αφορά την αρχή αυτή, χρησιμοποίησέ το ή θα το χάσεις. Είμαι αρκετά σκεπτικός σε σχέση με αυτό. Αυτή τη στιγμή οι δρόμοι αυτοί δεν υφίστανται καν, επομένως μιλάμε για πραγματική ζημία. Δεν υπάρχει καν η δυνατότητα χρησιμοποίησής τους. Σαφώς, ορισμένα κράτη-μέλη δεν μπορούν να αξιοποιήσουν τις ευκαιρίες που τους δίνονται από τα ευρωπαϊκά κονδύλια, από όλα αυτά τα προγράμματα. Γι' αυτό ακριβώ το λόγο λέω και εγώ στη γνωμοδότηση ότι θα πρέπει να αυξηθεί η ροή πληροφοριών που πηγαίνει προ τα κράτη-μέλη όσον αφορά τι δυνατότητε χρηματοδότηση. Θα ήθελα να ολοκληρώσω το σημείο αυτό και ελπίζω πραγματικά ότι θα καταθέσετε καλέ τροπολογίε που θα μα επιτρέψουν να έχουμε μια καλύτερη γνωμοδότηση. Ελπίζω να καταφέρω να τι ενσωματώσω όλε. Δεν νομίζω ότι υπάρχουν πολιτικέ αντιπαλότητε όσον αφορά το προσυζήτηση αυτό ζήτημα. Σα ευχαριστούμε κύριε Σιγητά, λέει η Πρόεδρο. Σα πενθυμίζω ότι η προθεσμία κατάθεση τροπολογιών είναι η 22 Φεβρουαρίου στι 6 το απόγευμα. Συνεχίζουμε τώρα με το επόμενο σημείο της ημερήσιας διάταξης που αφορά την απαλλαγή 2016, Γενικός Προπολογισμός Ευρωπαϊκής Ένωσης, Ευρωπαϊκή Επιτροπή και άλλοι οργανισμοί. Αρμόδια Επιτροπή είναι η Επιτροπή Ελέγχου του Προπολογισμού. Έχουμε εδώ πολλούς εισηγητές. Να δώσω καταρχά το λόγο στην κυρία Τεμόντε και έπειτα στον κύριο Φέρμπερ, τον κύριο Νταλούντε, την κυρία Μάισνερ και εν τέλει πάλι στην κυρία Τεμόντε, διότι είναι υπεύθυνη και για την ασφάλεια της αεροναυτιλίας με τον οργανισμό ΣΕΖΑΡ. Ξεκινάμε εσάς κυρία Τεμόντε, έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ πρόεδρε. Καταρχάς θα ήθελα να ευχαριστήσω τους και όδης και όλους τους συναδέλφους οι οποίοι κατέθεσαν τροπολογίες. Είναι 20 συνολικά οι τροπολογίες αυτές. Έχουμε καταφέρει να καταλήξουμε σε συμβαστικά κείμενα, πέρα από το κείμενο του σχεδίου γνωμοδότησης, στα πλαίσια, στα του οποίου συμφωνούμε όλοι ότι στα, με τα TEN-T έχουμε καταφέρει να πετύχουμε την ευκταία πρόοδο. Και γι' αυτό το λόγο, ω συντονιστέ, θέλουμε να υπάρχει μια καλύτερη αξιολόγηση των έργων εκείνων που έχουν ολοκληρωθεί και μια αξιοποίηση των βελτιώσεων που έχουν επέλθει και μια καλύτερη ανάλυση των ανισορροπιών και των ανισοτήτων που υπάρχουν μεταξύ των κρατών μελών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Απευθύνομαι εδώ πέρα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή αλλά και εδώ στις αρμόδιες αρχές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου λέγοντας ότι θα πρέπει να υπάρχει ένας μηχανισμός για να αυξηθεί η προστιθέμενη αξία των κοινοτικών κονδυλίων προκειμένου να ολοκληρωθούν τα δίκτυα TEN-T. Εν κατακλείδη λέμε ότι θα είναι πάρα πολύ σημαντικό να υπάρχει μία ενδελεχής ανάλυση όσον αφορά την αποτελεσματικότητα των κονδυλίων, να δούμε δηλαδή ποια είναι τα πραγματικά αποτελέσματα στα οποία οδηγούν και θα πρέπει και αφού να ληφθεί υπόψη στο μελλοντικό πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο. Αυτό το έχουν τονίσει και οι συνάδελφοι με τις τροπολογίες τους και λέμε επίση ότι θα είναι πάρα πολύ σημαντικό να υπάρχει απαραίτητη χρηματοδοτική και τεχνική στήριξη όσον αφορά το στόχο αυτό. Για άλλη μια φορά ευχαριστώ τους συναδέλφους για τη συνεισφορά τους. Ευχαριστούμε πολύ κυρία Ντεμόντε. Ο κύριος ε, Βιμ Βαντεκάμπ έχει το λόγο και αντικαθιστά τον κύριο Φέρμπερ. Ευχαριστώ πρόεδρε. Ο Μάρκος Φέρμπερ εξέτασε και τις δύο απαλλαγές. Και κατήρτισε μία έκταση, συζήτησε κάποιες τροπολογίες και κατά τα άλλα δεν υπάρχει οποιοδήποτε θέμα προς συζήτηση και μπορούμε αύριο να περάσουμε στην ψηφοφορία. Σας ευχαριστώ. Κύριε Βίμφαν Νικάμπ, ο κύριος Τελούντε έχει το λόγο. Ε, thank you, Chair. Ευχαριστώ, Πρόεδρε να εξηγήσω, να μιλήσω καταρχάς με τις τροπολογίες που λάβαμε. Λάβαμε σημαντικές τροπολογίες ό,τι αφορά την απάτη, το Brexit, την έρευνα, την καινοτομία. Ε, τις καλωσορίζουμε όλες αυτές τις τροπολογίες, εκτός από μία πιστεύουμε ότι θα, έχει, θα είναι σκόπιμο να κοιτάξουμε τον κανονισμό για το πόσο μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε το σωρευμένο πλεόνασμα για να υποστηρίξουμε σωστά τους πόρους μας. Δεν υποστηρίζουμε την τροπολογία 4 για τους ε, απαλλαγέ. Τώρα μιλώ εξ ονόματα του κυρίου Eichhout, όπου εστιαζόμαστε σε θέματα διαφάνεια. Και εδώ φυσικά είμαστε υπέρ σε ό,τι αφορά και την αποφατικότητα και την διαφάνεια. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Ντελούντα. Η κυρία Μέισνερ έχει το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Να μιλήσω για την ΕΜΖΑ. Η ΕΜΖΑ έκανε πολύ καλή δουλειά της, όπως είπα και την προηγούμενη φορά. σε ό,τι αφορά το προσωπικό, την αύξηση του προσωπικού που ήταν απαραίτητη, όλα είναι σωστά και ορθά. Κάναμε μόνο τέσσερις τροπολογίες λάβαμε και τις ε, συνενώσαμε σε μια συμβαστική πρόταση και νομίζω ότι και οι σκιώτες ήταν όλοι ικανοποιημένοι. Έχουμε συνεργές με, άλλα, με άλλες υπηρεσίες, σε ό,τι αφορά για παράδειγμα κυρίως το θέμα της προσφυγικής κρίσης και εδώ νομίζω ότι η ΕΜΖΑ έδρασε σωστά και άρα όλα καλά και ωραία. Ευχαριστούμε την κυρία Μέσνερ. Και η κυρία Ντεμόντα έχει πάλι το λόγο. Ευχαριστώ πρόεδρε και επ' αυτού θα πρέπει να συγχαρώ και να ευχαριστήσω τους συναδέλφους για τη συνεισφορά τους. Έχουμε μόνο 12 τροπολογίες χωρίς προβλήματα ε, και αυτό που θέλαμε ήταν να αποτιμήσουμε το κόστος καθώς και ορισμένες προβλέψεις για πολιετής συμβάσεις πριν από την διαδικασία διαγωνισμού. Νομίζω ότι όλοι συμμερίζονται αυτή την άποψη γιατί αυτός είναι ο κανόνας για όλους τους διαγωνισμούς. Άρα δεν υπάρχει θέμα για την ε, έγκριση του σχεδίου γνωμοδότησης. Ευχαριστούμε κυρία Ντεμόντε. Τώρα ανοίγουμε τη συζήτηση για το σύνολο των οργανισμών και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ο κύριος Λωτός ζήτησε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Συμφωνήσαμε ότι έχει επιτελεστεί πρόοδο σε σχέση με την υποστήριξη του ΤΕΝΤΗ από διαρθρωτικά ταμεία και από το Ταμείο Συνοχής. Χρειάζεται μεγαλύτερη αξιολόγηση για να δούμε ποια, ποιες είναι οι επιπτώσεις αυτών των ταμείων σε άλλες πολιτικές και αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να γίνει ένας γεωγραφικός καταμερισμός. Όμως δεν θα πρέπει να υπάρχει ξεχωριστή γραμμή του προϋπολογισμού για τον τουρισμό θα πρέπει να υπάρχει μία πρόσμιξη και θεωρούμε ότι χρειάζεται πραγματογνωμοσύνη για να έχουμε τα περισσότερα ευεργετήματα. Υποστηρίζουμε, υποστηρίζουμε λοιπόν την απαλλαγή για την ε, έμσα Θεωρούμε ότι μπορούμε να δεχτούμε τη γνωμοδότηση για τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Ασφάλειας στη Θάλασσα και αυτό αφορά και τον ε, ε, Οργανισμό για τους Σιδηροδρόμους. Ο κύριος Τέλιτσκα έχει το λόγο. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να μιλήσω για τον ε, προϋπολογισμό και όπως είπα την ε, ε, προηγούμενη φορά είναι πολύ καλή η πρόταση και χαίρομαι διότι οι τροπολογίες έχουν ένα θετικό αντίκτυπο και θεωρούμε ότι χρειάζεται μία συνολική αξιολόγηση όπως είπε και η κυρία Τεμόντε, θα πρέπει να δούμε ποιο είναι το προσδοκόμενο αποτέλεσμα. Τώρα, θα μιλήσω εξ ονόματος ε, του συναδέλφου Μίλτενμπουργκ για το ΣΥΖΑΡ και την ΕΑΖΑ από πλευράς ε, του δικού μας κοιόδους θα ήθελα να πω ότι δεχόμαστε την απαλλαγή για το ΣΥΖΑΡ ως προς την ΕΑΖΑ υπάρχει ένα αρνητικό πρόσημο στην τροπολογία 6. Θεωρούμε ότι θα πρέπει να υπάρχει ειδική ευρωπαϊκή νομοθεσία για τα drones και θα πρέπει να ε, λάβουμε υπόψη τροπολογία 7 που συνδυάζει και τις δύο συνιστώσεις. Θα θέλαμε επίσης να απαλληφθεί το τελευταίο μέρος της τροπολογίας 7 και στην τροπολογία 4 αρνούμεθα να υπάρξει μείωση της επιδότησης γιατί τα δύο τρίτα της ΕΑΣΑ καλύπτονται από, τις, από τη βιομηχανία. Αυτό αφορά και την πιστοποίηση προϊόντων. Όμως η, εποπτεία, η ρυθμιστική εποπτεία και το κόστος της δεν θα πρέπει να καταβάλλεται από τη βιομηχανία. Γι' αυτό θεωρώ ότι χρειάζεται η συνεισφορά του προϋπολογισμού, του κοινοτικού προϋπολογισμού και γι' αυτό έχουμε υποβάλει την τροπολογία υπαριθμών 4. Η κυρία Φώστερ. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κυρία Ντεμόντε για την εξαιρετική εργασία. Για την ΕΑΣΑ και το ΣΕΖΑΡ, καταρχήν ως προς το ΣΕΖΑΡ προσπαθούμε να αποστείλουμε ένα πιο δυνατό στεναρό μήνυμα προς τα κράτη-μέλη γιατί δεν μπορούμε να εφαρμόσουμε το δεύτερο σκέλος διότι υπάρχουν πολιτικοί περιορισμοί και ε, δεν υπάρχει πρόοδος ως προς τον ε, κατακαιρματισμό για την αεροναυτιλία, γιατί φυσικά ε, ανθίστανται τα κράτη-μέλη. Φυσικά θα υποστηρίξουμε την απαλλαγή. Επίσης αναγνωρίσουμε το θέμα των ε, μη επανδρομένων αεροσκαφών και θα υπάρξει μια επέκταση αυτής της δραστηριότητας για τα προσεχεία έτη. Ως προς την έκθεση Ντελούντε για την ΕΑΣΑ, συμφωνώ με τον κύριο Τελίτσκα για την τροπολογία 4. Ο προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης συνδράμει πολύ περιορισμένα. Γι' αυτό είτε θα κρατήσει αυτό το στάτους παρά το γεγονός ότι τα τρία τέταρτα του προϋπολογισμού της ε, καλύπτονται από τη βιομηχανία και εάν θέλουμε η Ευρωπαϊκή Ένωση να συμμετάσχει σε αυτό το επίπεδο, τότε η χρηματοδότηση θα πρέπει να διατηρηθεί. Καλωσορίζω την πρόταση για τη μεγαλύτερη εμβέλεια χρήσης των drones και έχω μία ερώτηση προς τον κύριο Ντελόντε στη τροπολογία 3 για την διαφοροποίηση με βάση τις θέσεις διοικητικές και μη. Ε, όμως συνολικά θα υποστηρίξουμε τις απαλλαγές. Απλώς θέλουμε να γίνουν ορισμένες ε, διασαφηνίσεις και ευχαριστούμε πολύ και την κυρία Ντεμόντ. Ευχαριστούμε πολύ κυρία Φώστερ. Ο κύριος Τεντενέσκι έχει το λόγο. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι μια κοινή επιχείρηση ε, Shift to Rail που αποτελεί την πιο νεόκοπη επιχείρηση η οποία όμως απέδειξε την αξία της και έχει και προοπτικές για το μέλλον. Έτσι μπορέσαμε να βελτιώσουμε τις σιδηροδρομικές ε, μεταφορές εκτιμώ την εργασία του συναδέλφου, του κυρίου Φέρμπερ, γιατί αποτελεί μία πολύ καλή βάση για την Επιτροπή μας και θεωρώ ότι με τις τροπολογίες ε, βελτιώθηκε το πλαίσιο του Shift to Rail. Χαίρομαι που ο κύριος Φέρπερ δέχτηκε τις τροπολογίες μου και θεωρώ ότι έτσι θα μπορέσουμε να λειτουργήσουμε καλύτερα στο μέλλον και θα βελτιωθούν και οι προοπτικές των σιδηροδρομικών μεταφορών μέσα στα πλαίσια των μεταφορών στην Ευρώπη. Τώρα θα ξαναδώσω το λόγο στον εισηγητή, στον κύριο Νταλούντε. Έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ. Όσον αφορά την τροπολογία παριθμών 3 από τους φιλελεύθερους, λέγεται εδώ πέρα ότι ε, υπάρχει μια διακριτική μεταχείριση ε, ή μάλλον μια, ένα χάσμα όσον αφορά τον τρόπο με τον οποίο διορίζονται κάποια μέλη του προσωπικού. Σε σχέση δηλαδή με την διάκριση που γίνεται μεταξύ AD και AST διαφορετική μεταχείριση σε σχέση με αυτό το οποίο προβλέπεται από άλλου οργανισμού. Την ερώτησή θα πρέπει όμω να απευθύνεται στου συντάκτε αυτή τη τροπολογία. Σα ευχαριστούμε, κυρία Ντεμόντ, έχει το λόγο. Σα ευχαριστώ. Παίρνω το λόγο μόνο σε σχέση με την ε, ΕΑΖΑ. Εμείς υποστηρίζουμε τις ε, τροπολογίες που έχουν υποβληθεί Θέλουμε δηλαδή να τονίσουμε ότι η γνωμοδότηση είναι πολύ καλή ποιότητα και το ίδιο ισχύει και για τι τροπολογίε με τι οποίε συμφωνούμε και τι οποίε στηρίζουμε. Ευχαριστούμε πολύ, κυρία Μάισνερα. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Δεν νομίζω ότι ακούστηκε κάποια ερώτηση για την ΕΜΣΑ, έτσι δεν είναι. Πολύ ωραία. Λοιπόν, θα ψηφίσουμε αύριο για τις απαλλαγές αυτές στις 9 ώρα το πρωί για το σύνολο των προτάσεων αυτών απαλλαγών όσον αφορά όλους τους οργανισμούς. Συνεχίζουμε τώρα με την Ευρωπαϊκή Στρατηγική για Συνεργατικά και Φυή Συστήματα Μεταφορών. Η συγκητής είναι ο κύριος Ουλεή. Έχετε το λόγο κύριε Σιγητά και έπειτα θα ακούσουμε τους σκιώδη συγκητές και έπειτα θα δούμε τι έχει να μας πει και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Κύριε Ουλεή, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Αξιότιμα μέλη της Επιτροπής Μεταφορών. Θα ήθελα καταρχάς να ευχαριστήσω και να συγχαρώ όλους τους συναδέλφους με τους οποίους συνεργάστηκα για την έκθεση αυτή. Να ευχαριστήσω επίσης και το προσωπικό της Γραμματείας και αναφέρομαι βέβαια στην γραμματεία της Επιτροπής μας και θα ήθελα όμως να συγχαρώ και τους σκιώδεις εισηγητές οι οποίοι έκαναν μια εξαιρετική δουλειά. Αγαπητοί συνάδελφοι, Έχω ασχοληθεί με διάφορε εκθέσει, αλλά πρώτη φορά βλέπω τόσο μεγάλο μέρο εργασία να γίνεται από του σκιώδει συγητέ. Προτού ψηφίσουμε την έκθεση αυτή, θα ήθελα να σας πω ότι ξεκινήσαμε περίπου πριν από ένα χρόνο να επεξεργαζόμαστε την έκθεση αυτή. Πέρασε περίπου λοιπόν ένα έτος, κατά τη διάρκεια του οποίου εκπονούσαμε την ε, έκθεση αυτή. Θα θυμάστε ότι υποβλήθηκε το Σεπτέμβριο, τη συζητήσαμε εν συνεχεία τον Νοέμβριο και κατατέθησαν τελικά 176 συνολικά τροπολογίες και ήρθαμε σε επαφή επίσης και με 17 εκπροσώπους από το βιομηχανικό κλάδο. 41 συμβαστικές τροπολογίες είναι το αποτέλεσμα τελικά των συζητήσεων που κάναμε. Συμφωνώ με τις περισσότερες από αυτές, καθώς επίσης και με την πλειοψηφία των πολιτικών ομάδων. Χρειάστηκε να κάνουμε περαιτέρω συζητήσεις για συγκεκριμένε μόνο τροπολογίες οι οποίες έχουν να κάνουν μάλλον με συγκεκριμένες προθεσμίες εφαρμογής συγκεκριμένων προγραμμάτων ή προθεσμίες οποίων θα για τις οποίες θα πρέπει να έχει προβλεφθεί μεγαλύτερη πρόοδος. Εγώ θα ήθελα να προχωρούσαμε λίγο πιο γρήγορα, αλλά από ό,τι φαίνεται δεν μπορούμε να ασκήσουμε εμεί ως Κοινοβούλιο άμεση πίεση σε άλλους εξωτερικούς ευρωπαϊκούς οργανισμούς. Ακόμα και όταν μιλάμε για κάποια πολύ σημαντικά ζητήματα, όπως αυτά τα οποία επεξεργαζόμαστε στην έκθεση αυτή και τα οποία επηρεάζουν ε, όλο τον πληθυσμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ε, όλους τους ανθρώπους, Ευρωπαίους πολίτες, από την πιο τρυφερή ως την πιο προχωρημένη ηλικία. Επίσης, ε, Έχουμε τρεις ε, επιτροπές, ENVI, IMCO και ΛΥΜΠΕ, οι οποίες γνωμοδοτούν και έχουμε καταφέρει να συμπεριλάβουμε ήδη στην ε, πρόταση έκθεσης ένα μεγάλο μέρος από τις προτάσεις τους. Θα ήθελα εγώ να αφαιρθώ τώρα σε κάποια σημεία επί την οποία έχει αλλάξει η διατύπωση χάρη στην συμβολή των σκιωδών εισηγητών. Οι σκιώδε ηγητέ προφανώ γνωρίζουν πληροφορίε αυτέ ήδη, οι υπόλοιποι συνάδελφοι όμω θεωρώ ότι θα πρέπει να ενημερωθούν. Αναφέρομαι καταρχά στην παράγραφο 15 όσον αφορά την τεχνολογική ουδετερότητα. Είναι ένα ζήτημα το οποίο συζητήσαμε εκτενέστατα. Είπαμε ότι θα πρέπει να παραμείνουμε ανοιχτοί, διαλλακτικοί απέναντι στι τεχνολογίε εκείνε οι οποίε ακόμα δεν έχουν αναπτυχθεί πλήρω ή απέναντι σε εκείνε οι οποίε θα εμφανιστούν στο μέλλον. Γι' αυτό το λόγο μιλάμε εδώ πέρα για ουδετερότητα της τεχνολογίας. Ξέρετε ότι ήδη αναφερόμαστε σε εφαρμογές που χρησιμοποιούνται σε εφή τηλέφωνα ή σε άλλες συσκευές. Είναι σημαντικό όμως να καταφέρουμε να προβλέψουμε και λίγο τι επιφυλάσσει το μέλλον σε σχέση με την τεχνολογία αν ε, αναφερόμασταν ε, πριν από μερικά χρόνια σε όλα αυτά τα οποία μπορούμε να κάνουμε τώρα με ένα κινητό τηλέφωνο, πάρα πολλοί θα μας λέγανε ότι όλα αυτά αποτελούν επιστημονική φαντασία. Παρ' όλα αυτά τώρα αποτελούν πραγματικότητα. Ας μην αποκλείουμε λοιπόν τις νέε αυτές τεχνολογίες αλλά και τις διαλειτουργικές τεχνολογίε, όλε εκείνε τι ε, πλατφόρμες CITS με τα 19 αυτά συμμετέχοντα μέλη τα οποία μπορούν να οδηγήσουν στο ITCSG5, τα νέα δηλαδή αυτά συστήματα τα οποία θα αρχίσουν συντομότατα να εφαρμόζονται. Χαίρομαι λοιπόν πάρα πολύ που υπάρχουν ήδη κάποια κρατημέλη, 19 το αριθμό, που έχουν ήδη προσχωρήσει στην πλατφόρμα αυτή. Πρέπει επίσης να σας πω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να υπάρχει η απαραίτητη συμβατότητα εκ των προτέρων και εκ των υστέρων και απαραίτητη διαλειτουργικότητα. Οι συμβαστικές προτάσεις αναφέρονται σε επικοινωνίες που βασίζονται σε δορυφόρους ή σε τεχνολογίες που βασίζονται στην κινητή τηλεφωνία. Επί των σημείων αυτών συμφωνήσαμε με τους υπόλοιπους σκιώδεις εισηγητές και αναφερόμαστε εδώ πέρα επίσης στην Συμβαστική 22 παράγραφος 20, ένα ζήτημα το οποίο συζητήσαμε εκτενέστατα με τους σκιώδεις εισηγητές. Συντοπίσαμε ότι το ζήτημα αυτό είναι πολύ σημαντικό Ορισμένοι είπαν ότι ενδεχομένω μετά όσα λέμε εδώ πέρα να ανοίγουμε το κουτί τη Πανδώρα και να αντιμετωπίσουμε πολλέ προκλήσει στο μέλλον. Παρ' όλα αυτά, νομίζω ότι όλοι συμφωνούμε ότι ε, τα δεδομένα τα οποία φέρουν τα οχήματα και η πρόσβαση στα οχήματα αυτά είναι πάρα πολύ σημαντικό ζήτημα. Ξέρετε ότι η ενταλλαγή των δεδομένων αυτών θα μας απασχολήσει και για τις οδικές μεταφορές αλλά και για πολλές άλλες μεταφορές. Έγιναν έντονες συζητήσεις και μια έντονη ανταλλαγή email για το ζήτημα αυτό και καταλήξαμε σε μια συμβαστική πρόταση. Καλούμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προχωρήσει συγκεκριμένε νομοθετικέ διατάξει μέχρι το τέλο του έτου. Παρ' όλα αυτά, θέλουμε εμεί να μπορούμε να ελέγχουμε ποιο και με ποιο τρόπο έχει πρόσβαση στα δεδομένα αυτά, τα on-board data, αυτά δηλαδή τα οποία αποθηκεύονται στα οχήματα. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους συναδέλφους εκείνους οι οποίοι συνέβαλαν πάρα πολύ σε όλες εκείνες τις τροπολογίες που έχουν να κάνουν με το σύστημα CITS. Συμφωνώ επίση με την τροπολογία 172. Κύριε Μιούτεμπερκ, αποστέλω και σε εσά ένα μήνυμα Ξέρετε εδώ πέρα ότι υπήρχε ένα αρνητικό πρόσημο στον κατάλογο των ψηφοφοριών. Ήταν λάθος προφανώ αυτό. Σαφώς είμαι υπέρ της τροπολογίας 172. Δεν υπάρχει λόγο λοιπόν να την συζητήσουμε περαιτέρω. Τονίζω, επαναλαμβάνω ότι και εγώ συμφωνώ με την τροπολογία αυτή. Συμβαστική 14. Τη συζητήσαμε και αυτή εκτενώ. Ο κύριο Μίτεμπερκ είχε πει ότι θα πρέπει να κατονομάσουμε εδώ πέρα τους ε, κατασκευαστές ε, οχημάτων, αυτοκινήτων. Έλεγε επίσης ότι δεν θα πρέπει να αποθηκεύουν τα δεδομένα των επιβατών στα αυτοκίνητα αυτά. Συμφωνώ με την ανησυχία αυτή, αλλά θα ήθελα και από αυτού να προτείνω μια συμβαστική πρόταση. Δηλαδή, να μπορεί ο οδηγός να δίνει εκ των προτέρων τη σύμφωνη γνώμη για τη χρησιμοποίηση του συστήματος e-call. Επίσης θα ήθελα να αναφερθώ και στις α, τροπολογίες του Αντιπροέδρου της Επιτροπής μας. Κάποιες τροπολογίες που κατατέθηκαν λίγο την τελευταία στιγμή στην τροπολογία 66 μπορώ να πω ότι συμφωνώ με το περιεχόμενό της. Χρησιμοποιείται όμως εδώ πέρα η φράση if appropriate. Δεν χρησιμοποιείται όμως η φράση αυτή στις υπόλοιπες τροπολογίες και νομίζω εδώ πέρα ότι θα πρέπει να έχουμε μια διατύπωση που να συμφωνεί περισσότερο με την προηγούμενη έκθεση, την έκθεση που είχαμε για το ζήτημα αυτό. Αγαπητοί συνάδελφοι, ήταν πραγματικά πολύ θετική και γεμάτη συζητήσει η περίοδο αυτή που προηγήθηκε, όλο αυτό το έτος το οποίο αναλώσαμε για την εκπόνηση έκθεση αυτή. Θα ήθελα λοιπόν να εγκρίνουμε την έκθεση αυτή αύριο για να καταφέρουμε τελικά να δημιουργήσουμε το σύστημα CITS. Ευχαριστούμε πολύ τον εισηγητή. Η κυρία Μπέρκινεν τώρα έχει το λόγο. Σα ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. σα ευχαριστώ πολύ και εσάς κύριε Σεγητά και όλους τους κοιότες. Να σας ευχαριστήσουμε όλους σας. Ε, νομίζω ότι οι Σεγητές οι συνεισηγητές μάλλον ε, κατέκτησαν ε, μια καλή βάση για την περαιτέρω δουλειά και νομίζω ότι μετά από τις διαπραγματεύσεις και τις τροπολογίες είναι ακόμα καλύτερη η έκθεση. Είναι καλή η συνεργασία και πολύ ισορροπημένο το αποτέλεσμα. Θα ήθελα να υπογραμμίσω τα ίδια στοιχεία όπως και ο εισηγητής. Και αυτά ασφαλώς ε, είναι και τα θέματα τα οποία μας απασχολούν στην έκθεση αυτή. Ένα από αυτά είναι η τεχνολογία, γιατί ξέρουμε ότι υπάρχουν διαφορετικές τεχνολογίες και φυσικά ότι η τεχνολογία διαρκώς αναπτύσσεται. Είναι πολύ λοιπόν σημαντικό να ε, συμφωνήσουμε σε μία προσέγγιση ιδιαίτερη ε, προς την τεχνολογία προκειμένου να έχουμε την τεχνολογία για τις βασικές αυτές ε, υπηρεσίες η ITA. Είναι σημαντικό να δώσουμε δυνατότητα πρόσβαση και ανταγωνισμού σε όλε τι τεχνολογίε, προκειμένου να υπάρχει και καινοτομία. Να υπάρχει δυνατότητα για καινοτομία. Αυτό λοιπόν θεωρώ ότι αποτελεί ένα πολύ καλό συμβιβασμό. Επίση, να τονίσω τη σημασία του συμβιβασμού υπερθυμών 22 γιατί είναι πρόσβαση σε δεδομένα εντό του οχήματο. Είναι σημαντικό λοιπόν όλη η αλυσίδα παραγωγή και ο τελικό χρήστη να μπορούν να επωφεληθούν από την ψηφιοποίηση. Γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει να υπάρχουν ίσοι α, όροι ανταγωνισμού και να προωθήσουμε και τις καινοτομίες. Εκ παραλληλού, είναι σημαντικό να υπάρχει και ασφάλεια σε ό,τι αφορά την πρόσβαση και την αποθηκεύση τέτοιων δεδομένων. Και άρα πιστεύω ότι είναι σημαντικό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να δημοσιεύσει μια νομισματική πρόταση, μια νομοθετική πρόταση για την πρόσβαση στα δεδομένα εντό του οχήματο ε, μέσα στο έτο το αργότερο. Αυτό είναι σημαντικό λοιπόν και είναι σημαντικό το κομμάτι τη έκθεση επί τη οποία έχουμε συμφωνήσει. Υποστηρίζουμε όλε τι τροπολογίε και θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε εκ νέου του συζητητέ ε, και του σκιώτε συζητητέ. Νομίζω ότι ήταν πραγματικά επικοδομητικέ οι συζητήσει, ανοιχτό πνεύμα για το συμβιβασμό και ήταν πραγματικά χαρά να συνεργαστούμε μαζί σα. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε την κυρία Μπερκανέν. Ο κύριος Σοντόσκι έχει τώρα το λόγο πάλι. Σας ευχαριστώ. Να ευχαριστήσουμε τον εισηγητή και εμείς για την πολύ καλή οργάνωση των διαπραγματεύσεων και να ευχαριστήσουμε και για τις συμβαστικές τροπολογίες. Υποστηρίζουμε όλες τις προσπάθειες που έχουν ως σκοπό τη δημιουργία ενός ευφυού συστήματος μεταφορών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πιστεύουμε ότι είναι ο μοναδικός τρόπος να μειωθεί ο ρυθμός των, οχημάτων, των ατυχημάτων στις ε, μεταφορές και να είναι οι μεταφορές πιο φιλικές πιο στο περιβάλλον. Ωστόσο, χρειαζόμαστε σαφές νομοθετικό πλαίσιο για να βοηθήσουμε τα κράτη-μέλη και τα σχετικά ερευνητικά ε, κέντρα. Η Ευρώπη λοιπόν θα πρέπει να αξιοποιήσει το πλήρες δυναμικό της για να μην ταλματώνει. Και χαίρομαι που συζητάμε συγκεκριμένες ημερομηνίε, συγκεκριμένα στοιχεία που θα πρέπει να κινητοποιήσουν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και αυτό είναι σημαντικό σε ό,τι αφορά τις μελλοντικές δημοσιονομικές προοπτικές που περιλαμβάνουν και τα φιλόδοξα σχέδια της ψηφιακής ατζέντα. Χωρίς τη σωστή υποστήριξη της έρευνας, της ανάπτυξης, την ανάπτυξη καινοτομία. Δεν μπορούμε να διανοηθούμε την ύπαρξη πρόοδου. Και υπάρχει και άλλο ένα σημαντικό θέμα. Το θέμα της προστασίας των δεδομένων και των προσωπικών δεδομένων και της προστασίας της ιδιωτικής σφαίρας. Αυτά τα στοιχεία, αυτά τα δεδομένα θα συλλέγονται και υπάρχει και ο κίνδυνος των κυβερνοεπιθέσεων. Αυτές είναι οι προκλήσεις που ελοχεύουν. Τα δεδομένα τα οποία συλλέγονται λοιπόν θα πρέπει δεν μπορούν να διακυβεύονται. Και κανένας κανονισμός δεν μπορεί να αποτελέσει εμπόδιο στην έρευνα σε ό,τι αφορά τη χρήση των βαλτίστων τεχνολογιών για να υπάρχει καλύτερη δυνατή επικοινωνία μεταξύ των ε, οχημάτων. Και χαίρομαι λοιπόν που αυτό αναφέρεται. Αναφέρεται στις τροπολογίες το θέμα της τεχνολογική ουδετερότητα. Η πολιτική ομάδα των συντηρητικών και μεταρρυθμιστών υποστηρίζει το κείμενο. Σα ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ο κ. Τελίντσικα τώρα έχει το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πολλά ακούσαμε ήδη και από του συναδέλφου ε, για την ε, έκθεση, για την καλή συνεργασία που υπήρχε με τον εισηγητή. Εγώ δεν μπορώ παρά να συμφωνήσω από πλευρά του κυρίου Φαν και σε ό,τι αφορά τη συνεργασία που ήταν καλή σε πολλά επίπεδα. Θα ήθελα να τονίσω ότι θα υποστηρίξουμε όλους ε, τους συμβιβασμούς τους οποίους πετύχαμε και καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή επίσης εξ ονόματος της ΑΛΔΕ να δημοσιεύσει νομοθετική πρόταση σε ό,τι αφορά την πρόσβαση των ε, δεδομένων εντό του οχήματο μέχρι το τέλο του χρόνου. Να συνάδει με τον κανονισμό για την προστασία των γενικών δεδομένων και πιστεύει ότι θα πρέπει να πετύχουμε τα πιο υψηλά πρότυπα προστασία του καταναλωτή. Συνολικά λοιπόν θεωρούμε ότι είναι μεγάλη σημασία του κειμένου και υποστηρίζουμε απόλυτα του συμβιβασμού. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κύριο Τελίνσκα. Ο κύριο Τελούντα έχει τώρα το λόγο. Ευχαριστώ πρόεδρε. Πολύ καλή έκθεση. Πολύ υποκοτομητική η διαδικασία συνεργασία. Ευχαριστούμε τον εισηγητή. Υποστηρίζουμε όλες τις συμβαστικές προτάσεις και την έκθεση στο σύνολό τη και σε ό,τι αφορά τις τροπολογίες για την διαλειτουργικότητα, την βιωσιμότητα, την προσβασιμότητα, ιδιωτική σφαίρα και προστασία δεδομένων, διαφάνεια. Όλα αυτά λοιπόν τα οποία είχαμε ζητήσει ενσωματώθηκαν και υποστηρίζουμε το κείμενο λοιπόν. Ευχαριστούμε λοιπόν ο κύριος Κόρ. Ευχαριστώ και από πλευρά μου να ευχαριστήσω τον εισηγητή για την πολύ καλή έκθεση. Πιστεύω ότι υπάρχει και έντονη σύνδεση με τη δική μου την έκθεση πρωτοβουλία ό,τι αφορά την προστασία των ανθρωπίνων ζωών στα, από ατυχήματα. Θα πρέπει λοιπόν να τα λάβουμε αυτή υπόψη. Σε ό,τι αφορά τη συμβαστική υπερθυμών 11, αναφέρεται ότι καλούμε, τονίζουμε ότι τα συστήματα θα πρέπει να συνεχίσουν να αναπτύσσονται και να ενσωματώνονται σε υποχρεωτική βάση. Δεν θέλουμε να είναι υποχρεωτικό αυτό για όλα τα συστήματα, μόνο για τα συστήματα ασφαλείας. Καλούμε να προσταθεί μάλλον λέξη certain driving assistance instruments και να συνεχίσει το κείμενο όσο έχει. Certain, να προσταθεί η λέξη certain, ορισμένα δηλαδή συστήματα, για να είναι και πιο συμβατό το κείμενο με το κείμενο της δικής μου έκθεσης, το οποίο εγκρίθηκε με μεγάλη πλειοψηφία. Ευχαριστούμε και να στραφούμε προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να δώσουμε το λόγο αν δεν είναι εδώ εκπρόσωπο τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ε, δεν μου αρέσει να περιμένω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ο κύριος Λύρη ίσως θα μπορέσει να απαντήσει τις ε, Α, κατέφθασε η Επιτροπή. Ο κύριος Βιμ Βαντεκάμπ πήγε να βρει την Επιτροπή, την οποία και βρήκε. Ε, έχετε το λόγο στην ε, έκθεση, για την έκθεση Λερή. Ο κύριος Βαντερλίντε. Όχι, όχι, ανταλλάξαμε ρόλους. Ωραία, η ομάδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ευχαριστώ και με συγχωρείτε που έφτασα, που φτάσαμε κάπως ε, αργά. Ε, επειδή πήρα βάρος στα Χριστούγεννα, αυτό δεν με κάνει και πιο γρήγορη. Εν πάση περιπτώσει, πέρα των αστεϊσμών, Είδαμε το σχέδιο γνωμοδότησης και την πολύ καλή εργασία που έχει γίνει από τα μέλη της Επιτροπής ε, με τις τροπολογίες, ε, κάτι το οποίο μας ενισχύει για να κάνουμε πολλά και πολύ γρηγορότερα και φυσικά να μπορέσουμε να χρησιμοποιήσουμε αυτή τη μεγάλη ικανότητα για τα συνεργατικά ευφυή συστήματα μεταφορών. Προσπαθήσαμε λοιπόν να προωθήσουμε μερικές αρχές, διότι αυτή η τεχνολογία ε, δεν είναι απομονωμένη, αφορά ε, μια ένα ευρύτερο συνεργατικό σχήμα κινητικότητας και υπάρχουν ε, και ιδιαίτερες πλατφόρμες που αφορούν όλα τα πλαίσια κινητικότητας μέχρι το 2031. άλλο σημαντικό σημείο που αφορά και τη γνωμοδότηση αφορά τις, το κατάλογο υπηρεσιών που θα αρχίσουν να ισχύουν από το 2019 και ε, ε, αναφερθήκαμε στους, ε, στις θαλάσσιες λεωφόρους έτσι ώστε να υπάρχει ένας διαλειτουργικός τρόπος λειτουργίας. Βεβαίως, πρόκειται για καθαρά τεχνολογικά σχήματα. Κάτι άλλο που θα ήθελα να τονίσω είναι το γεγονός ότι η ίδια η στρατηγική φτάνει σε ορισμένα ορόσημα ή στόχους. Βλέπουμε ότι η βιομηχανία είναι πολύ δραστήρια και προσπαθεί να τηρήσει την προθεσμία του 2019 και θεωρούμε ότι θα γίνει άμεση χρήση. Ένα άλλο θέμα είναι το θέμα της ε, κυβερνοασφάλειας. Υπάρχουν κατευθυντήριες γραμμές έτσι ώστε να υπάρχουν ε, κρυπτογραφημένα μηνύματα τα οποία να μπορεί, στα οποία να μην μπορεί κανείς να έχει πρόσβαση και να μην ε, μπορεί να τα ε, σπάσει χωρίς αυτό να αναστέλει τη διαλειτουργικότητα. Από πλευράς Επιτροπής λοιπόν προσπαθήσαμε να αρχίσουμε να αναπτύσσουμε την κατεξουσιοδότηση πράξη ε, CTS. Είχαμε συζητήσεις και με τη βιομηχανία. Το θέμα αυτό έχει οδηγήσει σε ιδιαίτερο ενδιαφέρον, σε εκδήλωση ενδιαφέροντος και νομίζω ότι ένα από τα σημεία που υποστηρίζουμε είναι η διαλειτουργικότητα ε, την οποία προωθεί και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έτσι ώστε να ενισχύσουμε τις επενδύσεις στον τομέα το ταχύτερο δυνατό βεβαίως ε, ε, μέσα στα πλαίσια της πλήρωσης όλων των προδιαγραφών ασφαλείας. Μίλησα και για την αρχή της ε, συμβατότητας καθώς και το έγγραφο στρατηγικής γιατί δεν στεκόμαστε στην βραχυπρόθεσμη στρατηγική. Προσπαθούμε να προωθήσουμε υπηρεσίες οι οποίες ε, να ε, έχουν να λάβουν υπόψη τις νέες εξελίξεις στο τομέα των επικοινωνιών, δυνατότητες 5G ε, μέσα στα πλαίσια των τηλεπικοινωνιών. Σε αυτό το στάδιο μπορώ να σας πω ότι υποστηρίζουμε την εργασία του Κοινοβουλίου και χαιρόμαστε για το ενδιαφέρον που έχει επιδείξει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Μέσα στα πλαίσια της εργασίας της Επιτροπής Μεταφορών. Ευχαριστούμε πολύ. Claire Ο συνάδελφος έχει κάτι να προσθέσει. Α, δεν έχει. Δίνω το λόγο στον εισηγητή. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Η εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ανέφερε ότι η Επιτροπή μας, η Επιτροπή Τραν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δείχνει ιδιαίτερα ενδιαφέρον για τη στρατηγική αυτή. Με εγώ σας υπόσχομαι ότι έτσι θα παραμείνουν τα πράγματα, θα συνεχίσουμε δηλαδή να εκδηλώνουμε ενδιαφέρον. Σας παρακαλώ πολύ λοιπόν, καλέστε μας σε όλους τους διαλόγους, σε όλες τις συναντήσεις και συνεδριάσεις που έχουν να κάνουν με το ζήτημα αυτό, με το CITS. Να ευχαριστήσω για άλλη μια φορά όλους τους συναδέλφους για τη συνεργασία τους και να πω δύο πράγματα ακόμα. Δέχομαι την πρόταση του Αντιπροέδρου μας, έχετε απόλυτο δίκιο, Όντως, θα πρέπει να εναρμονίσουμε τρόπον τεινά τις δύο εκθέσεις που έχουμε για το ζήτημα αυτό, πράγμα το οποίο σημαίνει ότι εμείς θα κάνουμε τις απαραίτητες τροποποιήσεις στη διατύπωση της έκθεσής μου, κανένα πρόβλημα προς αυτό. Και δεύτερον, θα ήθελα να καλέσω όλους τους σκιώδεις εισηγητές και συνεισηγητές να ξαναβρεθούμε και θα προσφέρω σε όλους σας ένα πολύ καλό μπουκάλι κρασί από την Ουγγαρία ήταν πολύ θετική συνεργασία που είχα μαζί σα. Ελπίζω ότι δεν θα έχουμε αύριο προβλήματα με τα μέσα μαζική μεταφορά και ότι θα είστε όλοι παρόντες στι 9 το πρωί για να υπερψηφίσουμε και να εγκρίνουμε αυτή την έκθεση. Σα ευχαριστώ πολύ. Σα ευχαριστούμε και εμεί, κύριε Σιγητά. Ελπίζω ότι οι σκιώδεις συγητές δεν θα κρατήσουν το μπουκάλι κρασί μόνο για τον εαυτό του, θα το μοιραστούν και με του υπόλοιπου. Πολύ ωραία. Ψηφίζουμε την έκθεση αυτή αύριο το πρωί από τι 9 και μετά. Λοιπόν, με λύπη σας λέω ότι ολοκληρώνεται στο σημείο αυτό η συνεδρίασή μας. Θα τα πούμε πάλι αύριο στις 9 το πρωί, αλλά οι στονιστές θα πρέπει να παραμείνουν στην αίθουσα, αλλά η συνεδρία των στονιστών θα ξεκινήσει σε 20 λεπτά, δηλαδή στις 40. 5 παρά 20 θα ξεκινήσει η συνεδρίαση των συντονιστών. Όλους οι υπόλοιπους θα σας δω αύριο το πρωί. Σας ευχαριστώ πολύ.